μια βούληση ε, ισχυρή ότι θα υπάρχει μια αυτόματη ε, διανομή των διαφόρων φυλαδίων των ενημερωτικών επιχάρτου ε, ώστε να υπάρχει καλή ενημέρωση. Σημεριζόμαστε την ανάγκη να συμπληρωθεί ο φάκελος αυτός. Ευχαριστώ πολύ. Ράιν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φιλελεύθερο συνάδελφο κύριο Κλίντς για την εξαίρετη εργασία του. Πραγματικά πιστεύω σε σύντομο χρόνο κατάφερε ο εισηγητής να βρει ένα καλό συμβασμό. Ακόμα και χωρί χρηματοπιστωτική κρίση είναι δύσκολα τα θέματα αυτά στο χειρισμό τους και στη διαχείριση γενικότερα. Τα γνωρίζω πολύ καλά διότι έχω εργαστεί σε αυτό το κλάδο στο ΟΣΕΚΑ ε, το 2001 είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί αποτελεσματικά η αγορά για τους επενδυτές, τους καταναλωτές. Και τελικά αυτό επιτυγχάνεται νομίζω. Θυμίζω ότι το 2001 η κατάσταση δεν ήταν καθόλου εύκολη και προφανής. Ήταν ακόμα πριν τη διαδικασία Λαμφαλουσί. Πολλά μέτρα ελήφθησαν τότε, αλλά χρειάζεται να ληφθούν και νέα. Είναι σημαντικό να ενισχύεται και η αγορά και η ασφάλεια των επενδυτών, αλλά και η εποπτεία των ε, ΟΣΕΚΑ. Το είπε και ο Επίτροπος ο ίδιος. Κύριε Πρόεδρε, ε, γίνεται μεγάλος λόγος για αυτό το ευαίσθητο και λεπτό θέμα του διαβατηρίου για τις εταιρείες διαχείρισης. Ακούσαμε διάφορα σχόλια, αλλά νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση. Είναι καλό να επιμένουμε πάντα στον ανταγωνισμό και στην εξωστρέφεια για να είναι αποτελεσματική μια αγορά και να λειτουργεί σωστά. Και επίσης να είναι καλές και πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές. Να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ποσότητα και την ποιότητα της πληροφορίας. Όταν κατακλείζεται κανείς από πληροφορίες δεν είναι αυτό κατά ανάγκη σωστό και καλό. Αλλά θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι οι επενδυτές για να ε, παίρνουν τις αποφάσεις τους με τα λόγου γνώσεως. Νομίζω ότι βρήκα μια καλή ισορροπία. Η Ευρώπη ε, προφανώς και χρειάζεται εδώ μια καλώς λειτουργούσα αγορά και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες πραγματικά γνωρίζουν επιτυχία και εκτός της Ευρώπης οι ευρωπαϊκές. Εποφεληθούμε από αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ράιαν για 1,5 λεπτό. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κλίντς, τον εισηγητή, για την εξαίρετη πραγματικά έκθεσή του. Εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να συμφωνήσουν όλοι στο συμβιβασμό και τον συγχαίρω γι' αυτό. Η αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής φέρει περισσότερη γραφειοκρατία και μεγάλο βάρος και φόρτο και ορισμένα κράτη-μέλη ανησυχούν. Αλλά από την άλλη νομίζω προστατεύει και τους επενδυτές και τους καταναλωτές. Όπως ήδη είπαν ε, προλαλήσαντες, μια ανοιχτή αγορά είναι ε, καλή εξέλιξη και θετική και όταν είναι καλά ρυθμισμένη λειτουργεί σωστά. Σήμερα οι χρηματακορές είναι τόσο αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες που χρειάζονται κοινοί κανόνες για ε, τον κλάδο αυτό που είναι πλέον παγκόσμιος στις ε, επενδύσεις. Όχι μόνο στην Ευρώπη δηλαδή, αλλά και παγκόσμια ισχύ. Είναι ε, πρωτοφανή φαινόμενα αυτά και θα πρέπει να συνεργαστούμε παγκόσμια για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μεγάλη ευκαιρία διότι εορτάζουμε τη δεκάτη επέτειο της έλευσης του ευρώ που δείχνει από μόνο του πόσο σημαντική είναι η οικονομική συνεργασία και πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χώρα μου η Ιρλανδία είναι μέλος της Ευρωζώνης. Το κοινό το ενιαίο νόμισμα προσέφερε σταθερότητα σε δύσκολους χαλεπούς καιρούς παγκόσμια ύφεση στη Ιρλανδία. Αν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη, δυστυχώ. Θα είχαμε σήμερα τη μοίρα της Ισλανδίας. Θέλω να πω στα μέλη του Συμφέν κυρίω εδώ ότι αν είχε περάσει το δικό του, τώρα δεν θα ήμασταν στο ευρώ που μας έλεγαν και τότε ότι ήταν οπισθοδρόμηση. Δεν θα ήμασταν στην ΟΝΕ και η οικονομική μας θέση πραγματικά θα ήταν σήμερα σε επίπεδο Ισλανδίας. Θέλω να πω σε εκείνους στην Ελλάδα που στρέφονται κατά της Ευρώπης και απορρίπτουν τη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, διαχέουν έτσι μεγάλη σύγχυση στα πνεύματα για τις ε, δεχόμενες επιπτώσεις θα πρέπει να σκεφτούν τι σημαίνει οικονομικά αυτό για την Ιρλανδία. Θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της λήψης των αποφάσεων στην Ευρώπη. Αυτό ε, το χρειάζεται και η Ευρώπη και η επιχειρήση και η οικονομία μας. Σε ευχαριστώ. Um, Ο κύριος Πέρβης για δύο λεπτά. Uh, ε, ευχαριστώ. Παρόλες τις αμφιγνωμίες σχετικά με τον κανονισμό για τις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κλπ. Τούτο εδώ το παράδειγμα είναι ένα καλό παράδειγμα κοινή λογική και μετρημένη ρύθμιση του κλάδου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Σκλίντ δούλεψαν όπω έπρεπε και ευχαρίστω θα υποστηρίξω την πρόταση. Τα ο ΣΕΚΑ είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικότερα για τη σκοτσέζικη οικονομία. Είναι σημαντικό μέσο επένδυσης για του επενδυτέ, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και στι Ηνωμένε Πολιτείε ε, υπάρχει το πρότυπο το οποίο εμπνέει και εμά. Ο κύριο Κλίντς περιέλαβε πολλά από τα σημεία που θεωρούσα εγώ σημαντικά όπως η διαφοροποίηση σε νέα επενδυτικά προϊόντα για παράδειγμα με επαρκή ε, επίπεδα ασφαλείας και κοινή λογικής και κυρίως πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος στην Ευρώπη. Πολλά από τα οσεκά μας είναι πολύ μικρά και κατακαιρματισμένα. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε συγχωνεύσεις των οσεκά αυτών. Εγώ θα ήθελα μάλιστα αυτό να προχωρήσει ακόμη περισσότερο έτσι ώστε οσεκά με διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους να μπορούν να συγχωνεύονται ευκολότερα και να προσφέρουν στον επενδυτή πλήρη προστασία και ενημέρωση για τις αλλαγές αυτές. Και τέλος το διαβατήριο διαχείρισης, το οποίο είναι πολύ σημαντική νέα διάταξη που θα επιτρέψει ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακος και αποτελεσματικότητα, μείωση της γραφειοκρατίας και αυτό βεβαίως είναι προς το συμφέρον του επενδυτού. Άρα η αναθεώρηση θα ωφελήσει τον κλάδο και πιο σημαντικό ακόμη θα αποτελέσει όφελος για τον αποταμιευτή και τον επενδυτή και μάλιστα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Άρα ευχαρίστως υποστηρίζω την, πρόταση του κυρίου, την έκθεση του κυρίου Κλίντς. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε Μπερές. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα για την εργασία σας, τη δέσμευσή σας και την διαπραγματευτική σας ικανότητα. Η ΟΣΕΚΑ είναι τρόπο να το σήμα κατά ε, των ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Είναι καλό εξαγωγικό προϊόν. Αλλά στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ανισορροπίες, διότι στο κλάδο αυτό έχουμε χώρες παραγωγούς, χώρες καταναλώτριες και διαφορετικές στρατηγικές λοιπόν. Ένα από του στόχου τη αναδιατύπωση οδηγία είναι να οργανώσουμε υπό τι συνθήκε αυτέ μια πραγματική σωστή λειτουργία τη ενιαία εσωτερική αγορά των ΟΣΕΚΑ. Έχω λοιπόν τα εξή ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, Κάτι που επανειλημμένα ακούστηκε αυτό το ζήτημα του διαβατηρίου διαχείρισης. Και άκουσα τον Επίτροπο να μας ε, λέει ότι φοβάται μήπως δεν προετοιμαστεί καλά αυτό το διαβατήριο. Μα αγαπητέ κύριε Επίτροπε, θα πρέπει κανείς να έχει τη βούληση να το προετοιμάσει. Και έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν τελείως αποφασισμένος προς την κατεύθυνση αυτή ο Επίτροπος και χαίρομαι για τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έτσι ώστε στην αδιατύπωση της οδηγίας αυτής να ε, υιοθετήσουμε δημιουργήσουμε ένα πραγματικό διαβατήριο διαχείριση που να επιτρέψει στην εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί υπό φυσιολογικέ συνθήκες. Δεύτερη παρατήρηση. Ε, τι γίνεται με την παρακράτηση. Για παράδειγμα, ε, στην αναθεώρηση της οδηγίας, ε, αν ε, υποχρεώνουμε τις ε, τράπεζες να παρακρατούν το 5% των τίτλοποιήσεων που κυκλοφορεί στην αγορά, θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα και με ίσους όρους, γιατί θα πρέπει οι ίδιοι κίνδυνοι να διέπονται από τους ίδιους κανόνες. Να υπάρχουν υποχρεώσεις παρακράτησης και εκεί. Τρίτον, τι γίνεται με την εποπτεία. Κανείς εδώ δεν αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητά μας ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της εποπτείας. Όλοι περιμένουμε κατ' πρωτοβουλίας ε, του κυρίου ε, Παρόσο τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας Ζακ Ντελαρούσια. Αλλά έχει έτσι η κατάσταση που δεν μπορούμε να περιμένουμε επάπειρο ε, τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των συμπερασμάτων. Και θα πρέπει αυτό να έχει αντίκτυπο και στην εποπτεία μεταξύ των διαφόρων φορέων παραγωγών καταναλωτών ως ΕΚΑ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το διακύβευμα της εποπτείας εκεί. Και τελευταία παρατήρηση έχει να κάνει με τα φορολογικά ζητήματα και διακυβεύματα, τα είπε και ο εισηγητής και ο Επίτροπος δεσμεύτηκε. Τι κρύβεται πίσω από τα φορολογικά. Ε, ε, συγκαλισμένος προστατευτισμός και θα πρέπει και να το καταγγελμα αυτό αλλά και να το ξεπεράσουμε. Πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει ε, πρωτοβουλίε έτσι ώστε και στους ΟΣΕΚΑ η φορολόγηση να επιτρέπει ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών χωρί πρόσθετα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Σταρκεβιτσούτε για ένα λεπτό. Ήθελα να πω και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, ο οποίος μπόρεσε να βρει τον καλό συμβιβασμό. Δεν είμαι όμως πλήρως ικανοποιημένος με αυτήν την έκθεση. Πρώτον, επειδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ετοιμάσουν όλη την νομοθεσία ε, στην γλώσσα η οποία είναι η συνήθις. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι στα αγγλικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μειώσουμε την εργασία, την γραφειοκρατική των επενδυτικών ε, εταιριών. Αλλά δεν πρέπει να δώσουμε προτίμηση σε μία γλώσσα, να χρησιμοποιείται μόνο μία γλώσσα. Επιπλέον πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε επιπλέον νομική αβεβαιότητα, πάντως χάρη σε ποια γλώσσα θα δίνουμε ε, πληροφορίες στον καταναλωτή. Πώς θα τον ενημερώνουμε Πιστεύω ότι η ευθύνη, η εταιρική και οι όροι του ανταγωνισμού θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το να έχει κανείς ένα αποτελεσματικό σύστημα αυτός θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Εφόσον υπάρχει ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι δυνατόν να μειωθεί το κόστος για τους επενδυτές και συμφωνώ με τον εισηγητή για τα όσα λέει σχετικά με τις υφιστάμενες προοπτικές. Ε, που θα πρέπει να αντικατασταθούν με ένα έγγραφο το οποίο θα παρέχει σαφείς πληροφορίες στον δυνητικό, στον ενδεχόμενο επενδυτή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στην φορολογία. Πιστεύω ότι η πρακτική ε, εφαρμογή ε, του διαβατηρίου διαχείρισης μπορεί να καταστήσει ε, δύνατον τα χαρτοφυλάκια αυτά ε, να γίνουν διαθέσιμα σε όλη την κοινότητα και αυτό έτσι θα επιτρέψει να καλύψουμε τα κενά ε, στην αγορά. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Εκτιμώ την εργασία που κάνει το Κοινοβούλιο αυτό παρατηρήθηκε εδώ σε όλες ε, τις παρατηρήσεις. Δεν είναι βεβαίως ε, το τέλος της ιστορίας. Πολλά πρέπει να γίνουν ε, στα κρατη που θα έχουν το έργο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας και μέχρι το καλοκαίρι του 2011 θα πρέπει επίσης να υπάρξουν και οι εθνικοί ελεγκτές και επόπτες για την καλή εφαρμογή του διαβατηρίου. Θα πρέπει να διευκολυνθεί αυτή η εργασία στον τομέα αυτόν τον επενδυτικό της κοινότητας. Τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Κλίνς για δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και να συμφωνήσω μαζί του ότι όντως δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Ένα λόγος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο έχουμε επιβάλει σύντομες προθεσμίες είναι για να διασφαλίσουμε ότι πράγματι η εφαρμογή δεν θα καθυστερήσει αλλά ότι θα συνεχίσει με ταχύ ρυθμό γιατί βλέπουμε τις αγορές να αλλάζουν, να, αλλάζουν, να τροποποιούνται με ρυθμό καλπασμού. Η σημερινή συζήτηση έδειξε μια διακομματική υποστήριξη υπέρ της ε, συμβαστικής προτάσεως. Εγώ δέχομαι την άποψη της κυρίας Λούλινγκ που είναι κάπως διαφορετική. Είμαι ωστόσο πεπισμένος ότι το μέλλον θα δείξει ότι οι ανησυχίες της, της κυρίας Λούλινγκ δηλαδή ότι ε, το Λουξεμβούργο ως κέντρο ε, χρηματοπιστωτικών ε, δραστηριοτήτων θα χάσει σημασία δεν θα, δεν είναι δικαιολογημένη η ανησυχία αυτή. κυρία ε, Μπερές εξάλλου έχει δίκιο που λέει ότι πρόκειται πραγματικά για προσπάθεια δημιουργίας της ενιαίας αγοράς και στον τομέα των ε, ΟΣΕΚΑ. Μιλούμε για ενιαία αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη δεν υπάρχει ακόμη αυτή η ενιαία αγορά. Προχωρούμε σε μια νέα και πολύ φιλόδοξη συνεργασία των οργάνων αυτών. Και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, Αλλά πρέπει αυτά τα όργανα να μπορούν να συνεργαστούν και σε άλλους τομείς με τρόπο που να προκαλεί εμπιστοσύνη. Και εάν η οδηγία ασκήσει κάποια πίεση ε, προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο το καλύτερο. Τα ε, μέτρα τα οποία έχει αναφέρει ήδη ο Επίτροπος είναι πολλά και πρέπει να ε, προωθηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι αυτό είναι αλήθεια. Ο ίδιος ο κλάδος ωστόσο πρέπει να κάνει, να εκτελέσει τα καθήκοντά του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν έχουμε θίξει το θέμα του fund processing διότι αναμένουμε ότι ο κλάδος θα τηρήσει την υπόσχεσή του να ε, ρυθμίσει τα θέματα αυτά από μόνος του χωρίς εξωτερική νομοθετική πίεση. Ελπίζω σύντομα να ανταποκριθεί ή δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι στο ορατό μέλλον να αναλάβουμε δράση. Εν τέλει, επιθυμώ να ευχαριστήσω όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ιδίω το Συμβούλιο για την συνεργασία και την υποστήριξη, καθώ και του εκπροσώπους των άλλων κομμάτων, και ιδίω την κυρία Μπερέ, την κυρία Γκοτάρντι και τον κύριο Γκοζέ, αλλά και την Άστιτ Λούλινγκ, η οποία με το μαχητικό πνεύμα που την διακρίνει τοποθετήθηκε και σήμερα ε, προς υποστήριξη των ε, συμφερόντων της χώρας της. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 10.